Dear colleagues, can we start? Παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι να ξεκινήσουμε. Σας καλωσορίζω. Θα περάσουμε στις ψηφοφορίες, οπότε παρακαλώ να έχετε έτοιμες τις ε, κάρτες για την ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε το σχέδιο έκθεσης την παρακολούθηση της εφαρμογής ε, της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2016. Συμβαστική 1. Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται φεμ β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 όχι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 κατά αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ για να είμαστε βέβαιοι. Εγκρίνονται. Εσείς ψηφίσατε υπέρ ή κατά. Θέλετε να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Αλλά ήταν ούτως ή άλλως 12 προς 8. Το αποτέλεσμα άρα ήταν ξεκάθαρο. Εγκρίνονται λοιπόν. NV1 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. NV11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 5 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 5 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Αύκο 7 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ένβι 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αύκο 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε την Αύκο 6 παρακαλώ. Too many EPPs. Από το ΕΛΚ είστε υπεράριθμοι. εγκρίνεται. Πού είμαστε? Α, στην 39. Τροπολία 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Φεμ 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται ένβι 8 υπέρ κατά αποχές εγώ νομίζω εγκρίθηκα και για να το ελέγξουμε καλύτερα. Yes. Adopted. Εγκρίνεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβεβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ α καταπίπτει λάθος μου συγγνώμη 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 10 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. εγκρίνεται 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 5 7 υπέρ, καταπίπτει, καταπίπτει, λάθος μου. 5 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 5 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές, ένβ NV18 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε παρακαλώ την ένβ 18 Yes. It has been rejected. Απορρίφθηκε. Πηγαίνουμε στην 61. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Την 61. Εγκρίνεται με σαφή διαφορά. Λάθος μου. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική. Συμβιβαστική 13 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 14 Α, όχι, λάθος μου. Πρέπει να πάμε στην 65 υπέρ. Against. Κατά. Αποχές. Παρακαλώ, επαναλαμβάνω την ψηφοφορία. Υπέρ της 65. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ. Α, πρέπει να γίνει με ονομαστική κλίση, έχετε δίκιο. Άρχεται η ψηφοφορία. εγκρίνεται. Τροπολογία 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Πραγματικό συμβιβασμός. Να ελέγξουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 16 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 78 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 82 υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ την 82. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 88. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε την 88. Απορρίπτεται. 87 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 89 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αύκο 8 υπέρ, κατά, αποχές, συγγνώμη θα ήθελα να ελέγξουμε. Αύκο 8. Εγκρίνεται. Αύκο 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται.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 κατά αποχές εγκρίνονται 5-10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5-18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Αύκο 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ. Αύκο 14. Απορρίφθηκε. Φέμ 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται σχέδιο. Έκθεση συνολικά. Ψηφίζουμε με ονομαστική κλίση. ψηφοφορία. Από το ΕΛΚ είστε παραπάνω. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε το σχέδιο έκθεσης και συγχαρητήρια στον κύριο Ράντεφ. Α, συγγνώμη, στον κύριο Χρυσόγονο συγχαρητήρια. Και τώρα έχουμε την αναδιατύπωση για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Ονομαστικά θα ψηφίσουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια για κυρία Γκέριγκερ. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τις ψηφοφορίες. That's it, yeah? okay. so, now... Λοιπόν, τώρα να πάμε στο σημείο 1, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Να σας ενημερώσω ότι τα σημεία 3, 4, 12 και 15 αναβάλλονται. Το σημείο 11 θα συζητηθεί μετά από το σημείο 12. Το σημείο 13 θα συζητηθεί μετά από το σημείο 6. Το σημείο 19 θα συζητηθεί μετά από το σημείο 13. Αντιρρήσεις, όχι, επομένως εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να ζητήσω ε, να κάνετε λίγη ησυχία. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε με το σημείο 13, πληροφορίες για τη διαπραγμάτευση των μέσων εφαρμογής των διακανονισμών στην UN Central Και έχουμε εδώ εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας ενημερώσει. Να δώσω λοιπόν τον λόγο στην Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που πήρατε την πρωτοβουλία να οργανώσετε αυτή την ενημέρωση για τις διαπραγματεύσεις αυτές που είναι σε εξέλιξη. Λέγομαι Νόρ Χόφμερ, είμαι στη Γενική Διεύθυνση Justice της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ασχολούμαι με αυτές τις διαπραγματεύσεις εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχάς θα ξεκινήσω με ένα σύντομο ιστορικό αυτών των διαπραγματεύσεων στην 48η συνεδρία το 2015, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, η UNCTRAL, αποφάσισε ότι η ομάδα εργασίας 2, ε, η οποία συνήθως ασχολείται με την επίλυση διαφορών, θα πρέπει να ξεκινήσει εργασίες για το, το θέμα της εφαρμογής ε, των συμφωνιών διακανονισμών για να δει τις πιθανές ε, λύσεις και την πιθανή προετοιμασία ίσως και μιας ε, διάσκεψης ε, διατάξεις ε, πρότυπο ή διατάξεις νομοθετικές ή και κατευθυντήρες γραμμές. Το έργο της UN Central θέλει να προχωρήσει από τα θεμόλια που έχουμε το 2002 για το πρότυπο νόμο για τη συνδιαλλαγή, ώστε να υπάρχουν δυνατότητες διαπραγμάτευσης και επίλυσης διαφορών ε, διεθνώς μέσω ε, συμφωνιών και διακανονισμών οι πολυμερείς διεθνείς διαπραγματεύσεις για μια σύμβαση και ένα πρότυπο νόμο έχουν στόχο να υπάρχουν δυνατότητες διεθνών διακανονισμών, συνεχίζονται αυτές οι διαπραγματεύσεις και ε, ελπίζουμε να ολοκληρωθούν στα πλαίσια της Trail. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύεται αυτά τα μέσα εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει και της διαπραγματευτικής εντολής που της δόθηκε από το Συμβούλιο. Μέχρι τώρα έχουν γίνει έξι γύροι διαπραγματεύσεων. Ο τελευταίος γύρος έγινε το Φεβρουάριο του 2018 και υπήρξε γενική συμφωνία για το κείμενο του μελλοντικού μέσου. Θα έχουμε μία σύμβαση και ένα παράλληλο πρότυπο νόμου. Τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντανακλώνται πολύ καλά στο συμφωνημένο κείμενο. Όσον αφορά ε, τη διαδικασία για την έγκριση αυτών των μέσων σε διεθνές επίπεδο, τα μέσα θα παρουσιαστούν πλέον προς έγκριση στο ε, διοικητικό ε, συμβούλιο της Σιτράλ, που είναι η Επιτροπή της Σιτράλ στην ε, επόμενη σύνοδο του φορέα αυτού, του οργάνου αυτού, που θα γίνει τον επόμενο μήνα και εάν εγκριθούν τα μέσα θα υπάρξει από εκεί και πέρα και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στο δεύτερο εξάμεινο του 2018. Τώρα, δύο λόγια για τη γενική δομή των μελλοντικών μέσων. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, ε, τα μέσα θα καλύπτουν και την εφαρμογή των διακανονισμών και ε, τη διαδικασία βάσει της οποίας ο διακανονισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, για να αποδείξουμε ότι έχει επιληθεί η διαφορά. Τα μέσα αφορούν ε, διεθνείς εμπορικούς διακανονισμούς, επομένως ε, δεν ισχύουν ε, για αστικές ε, διευθετήσεις διαφορών, ε, ως αποτέλεσμα διαμεσολάβησης και αποκλείονται καταναλωτικά, οικογενειακά και θέματα κληρονομικού δικαίου. Η διαμεσολάβηση σε αυτή την περίπτωση θεωρείται μια διαδικασία στην οποία οι δύο πλευρές προσπαθούν να επιλύσουν τη διαφορά τους με φιλικό τρόπο με τη βοήθεια κάποιου τρίτου ή κάποιων τρίτων, των διαμεσολαβητών βεβαίως, οι οποίοι όμως ε, δεν έχουν την εξουσία να επιβάλλουν μία λύση στις δύο πλευρές. Αυτή είναι και η βασική διαφορά μεταξύ της διαμεσολάβησης και ε, μιας δικαστικής διαδικασίας τα μέσα δεν ισχύουν για δικαστική επίλυση διαφορών που είναι ε, ε, ε, διαδικασίες οι οποίες εγκρίνονται από το δικαστήριο ή γίνονται ενώπιον δικαστηρίου και επίσης δεν ισχύουν για διατησία. Και ο λόγος για τον οποίο εξαιρούνται αυτές οι διαδικασίες είναι γιατί αυτές οι μορφές διακανονισμών καλύπτονται από άλλα διεθνή μέσα, στην περίπτωση της δικαστικής επίλυσης διαφοράς από την ε, σύμβαση της Χάγης το 2005 για την επιλογή δικαστηρίου που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ε, μελλοντική σύμβαση για τις ε, αποφάσεις της Χάγης η οποία είναι υποδιαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή για το Διεθνές Δίκαιο και θα θυμάστε ότι έγινε και σχετική ακρόαση στην Επιτροπή σας πριν από δύο εβδομάδες αν δεν κάνω λάθος όσον αφορά τη διαδικασία της διαιτησίας ε, εξαιρούνται γιατί καλύπτονται από άλλα διεθνή μέσα, πιο συγκεκριμένα τη σύμβαση του 1958 της Νέας Υόρκης για την αναγνώριση ε, των ε, διαιτητικών αποφάσεων. Όσον αφορά το σύστημα εφαρμογής, αυτό είναι σχεδιασμένο για να υπάρχει μια διαδικασία η οποία θα διεξάγεται από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα στην οποία ε, υπάρχει εφαρμογή. Αυτή θα καθορίζεται από τον κανονισμό της χώρας ε, στην οποία γίνεται η εφαρμογή και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να πρόκειται για δικαστική αρχή, παρά το γεγονός ότι κάποιες χώρες μπορεί μέσω της διαδικασίας τους να καθορίσουν άλλη αρμόδια αρχή για αυτό το σκοπό, παραδείγματο χάρη ε, συμβολογραφική αρχή. Αυτός ο έλεγχος θα βασίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία καθορίζονται σαφέστατα στα μέσα. Το σύστημα ε, αυτό ε, χωρίζεται σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα είναι για ε, ενστάσεις οποίες θα πρέπει να παρουσιάσει η πλευρά η οποία είναι κατά τις εφαρμογές και θα περιλαμβάνουν κάποια στοιχεία όσον αφορά το διακανονισμό ή το γεγονός ότι ο διακανονισμός μπορεί να μην είναι οριστικός ή να μην είναι δεσμευτικός. Επιπλέον, μία συμφωνία διακανονισμού μπορεί να ε, μην εφαρμόζεται αν ο διαμεσολαβητής ε, παραβίασε τα πρότυπα τα οποία ισχύουν για αυτόν ή τη διαδικασία της διαμεσολάβησης ή ε, δεν παρουσίασε κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί να ήταν εις βάρος της αμεροληψίας τους ή της ανεξαρτησίας του. Η άλλη πλευρά, η άλλη ομάδα είναι αυτά τα οποία ισχύουν εξοφίκιο από την αρμόδια αρχή και αφορούν ε, παραβίαση της ε, δημόσιας πολιτικής στη χώρα στην οποία ζητάται η εφαρμογή ή εάν ε, το θέμα της διαφοράς δεν μπορεί να επιληθεί μέσω διαμεσολάβησης βαση δικαίου της χώρας. Επίσης υπάρχει δυνατότητα να, το ένα από τα συμβαλόμενα μέρη να κάνει μία δήλωση ότι η σύμβαση θα ισχύει μόνο στο βαθμό που οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για την εφαρμογή της σύμβασης. Το σχέδιο σύμβασης θα περιλαμβάνει επίσης και ε, μία ρήτρα για έναν περιφερειακό οικονομικό οργανισμό ολοκλήρωσης για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους όσον αφορά τα θέματα της σύμβασης. Το σχέδιο της σύμβασης περιλαμβάνει και το λεγόμενο, τη λεγόμενη ρήτρα αποσύνδεση του Περιφερειακού Οικονομικού Οργανισμού Ολοκλήρωση, που θα επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση προσχώρηση να ε, εφαρμόσει ε, κανόνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι ε, είναι επίμαχοι σε αυτέ τι περιπτώσει. Ε, ε, σύμβαση, αν εγκριθεί από τη UN Citral και μετά εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, κατά πάσα πιθανότητα θα τεθεί σε εφαρμογή το πρώτο εξάμεινο του 2019. Η σύμβαση θα τεθεί σε εφαρμογή έξι μήνες μετά από την ε, κατάθεση του τρίτου μέσου κύρωσης και όπως σας είπα υπάρχουν δύο παράλληλα μέσα. Το ένα είναι η σύμβαση και το άλλο είναι ε, το πρότυπο νόμου. Το πρότυπο νόμου θα συμπληρώσει λοιπόν ε, το κείμενο μοντέλο που υπάρχει του 2002 και επομένως θα υπάρχει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο το οποίο θα αφορά την εφαρμογή των διακανονισμών και ε, το κεφάλαιο αυτό θα περιλαμβάνει σχεδόν αντίστοιχες διατάξεις από αυτές, ε, με αυτές που μόλις σας περιέγραψα για τη σύμβαση. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, sir, for this presentation. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στα μέλη του, της Επιτροπής που είναι παρόντα. Έχετε κάποια σχόλια, κάποια παρατήρηση, παρακαλώ. Από ό,τι βλέπω δεν έχετε. Άρα ήταν πολύ εξαντλητική η παρουσίαση γιατί εξάντλησε όλα τα θέματα και όχι εμάς βεβαίως. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι έχουμε ολοκληρώσει την εξέταση αυτού του ζητήματος της ημερήσιας διάταξης. Μπορούμε επίσης να ευχαριστήσουμε θερμά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να προχωρήσουμε στο σημείο 19 ανταλλαγή απόψεων. Υπάρχει το εξής πρόβλημα. Αποουσιάζει ο εισηγητής για το σημείο 19 διότι έχει προγραμματιστεί η εξέταση του σημείου αυτού για τις 11. Άρα μας αναγκάζει η κατάσταση να κάνουμε διάλειμμα για καφέ, χωρίς να το επιθυμούμε. Επομένως, διακόπτουμε για καφέ και θα συναντηθούμε σε 20 λεπτά στις 11 ακριβώς. Ευχαριστώ. La commission de la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

Υπότιτλοι AUTHORWAVE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

Thank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

Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε ή να συνεχίσουμε. Είναι πιο σωστό να πω να συνεχίσουμε με την εξέταση του θέματος 19 στην ημερήσια διάταξη. Ανταλλαγή απόψεων για τις διαφανείς και με συνθήκες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγητής είναι ο κύριος Κώστας Χρυσόγονος και του δίνω αμέσως το λόγο. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα τελευταία 25 χρόνια η ευελιξία με τις νέες μορφές απασχόλησης ήταν βασικός μοχλός για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Από το 2014 έχουν δημιουργηθεί πάνω από 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 20% αυτών βρίσκονται σε νέες μορφές απασχόλησης. Η προσαρμοστικότητα των νέων μορφών απασχόλησης στις αλλαγές στο κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο επέτρεψε στα νέα επιχειρηματικά μοντέλα να αναπτυχθούν. Ωστόσο, οι τάσεις αυτές οδηγούν και σε αστάθεια και σε αυξημένη απουσία προβλεψιμότητα σε ορισμένες εργασιακές θέσεις, ειδικότερα για τους εργαζόμενους στις πιο επισφαλείς θέσεις εργασίας. Έχουμε μη κατάλληλα νομικά πλαίσια τα οποία μπορούν να επιβάλλουν στους ε, ε, εργαζόμενους να εργάζονται με μη σαφείς και άδικες πρακτικές σε μη σαφή εργασιακά περιβάλλοντα και έτσι είναι πολύ δύσκολο να ασκήσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα. Είναι 4 με 6 εκατομμύρια εργαζόμενα, ε, εργαζόμενοι απασχολούνται σε συμβάσεις με, ε, οι οποίες διακόπτονται, οι οποίες με την ημέρα, με την ώρα, οι οποίες είναι αβέβαιες και δεν μπορούν να εργαστούν από την άλλη για άλλο ε, εργοδότη, γιατί έχουν ειδικέ ρήτρε. Το 1 τέταρτο των προσωρινών, απασχολούμενων πηγαίνουν σε ε, μόνιμη θέση εργασίας και 28% αυτών που δουλεύουν προσωρινά αλλά επιθυμούν μόνιμη θέση εργασίας ε, το 2016 ε, έτσι είναι το ποσοστό αυτών που δουλεύουν προσωρινά από ανάγκη και όχι από επιλογή. Ορισμένα κρατημέλη έχουν υιοθετήσει νέες ε, νομοθεσίες, νέες κανονιστικές διατάξεις, έχουν αναπτυχθεί νέες συλλογικέ συμβάσεις εργασίας και έχουμε όλο και πιο αποκλίνοντα μεταξύ τους κανονιστικά και ρυθμιστικά συστήματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως αυξάνεται ο κίνδυνος ανταγωνισμού, διότι σε μια χώρα θα γίνεται undercutting, θα μειώνονται δηλαδή τα κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα και θα καθίσταται η χώρα πιο ανταγωνιστική. Είναι μη βιώσιμη αυτή η ανταγωνιστική πίεση για τα κράτη-μέλη, τα οποία έτσι δεν έχουν αρκετές εισπράξεις από το φόρο, δεν έχουν αρκετά έσοδα για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και συνεισφοράς, γιατί υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός με τη μείωση εργασιακών συνδικών και εργασιακών προτύπων στη διπλανή χώρα. Πρέπει να έχουμε επαρκή προστασία όλων των εργαζομένων και αυτό διασφαλίζει μεγάλα ωφέλη και κέρδη στην παραγωγικότητα για τους εργοδότες σε βάθος χρόνου και υπάρχει σύγκληση σε προς καλύτερες συνθήκες ζωής, βιωτικό επίπεδο και καλύτερες συνθήκες εργασίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι γνωστά. Για να τα λύσουμε και να έχουμε ένα βασικό επίπεδο ε, ε, συνολικής προστασίας στις μελλοντικέ συμβάσει απασχόλησης αλλά και στις υφιστάμενες, γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προτείνει τη σχετική οδηγία και είναι μία από τις βασικές έννοιες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να, σε συνέχεια του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων που δημιουργήθηκε. Και η προτινόμενη οδηγία θα πρέπει να καθορίζει ποιο είναι το παράνομο πλαίσιο και ποιο είναι το νομικό πλαίσιο για να μπορούμε να έχουμε εξέλιξη των προσαρμοστικών μορφών απασχόλησης. Γενικότερο πλαίσιο είναι να προωθήσουμε απασχόληση πιο ασφαλή, πιο προβλέψιμη να διασφαλίσουμε την προσαρμοστικότητα στην αγορά εργασίας, αυτό ναι, αλλά να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας και ε, το βιωτικό επίπεδο, τις συνθήκες ζωής. Συγκεκριμένοι στόχοι της οδηγίας είναι οι εξής. Πρώτον, να βελτιώσουμε την πρόσβαση των εργαζομένων στην πληροφόρηση σε σχέση με τις συνθήκες εργασίας τους. Δεύτερον, να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας για όλους τους απασχολούμενους, για όλους τους εργαζόμενους, ειδικότερα σε αυτούς που εργάζονται σε νέες μορφές απασχόλησης ή σε μορφές απασχόλησης που δεν ε, μπαίνουν σε κάποια συγκεκριμένα πρότυπα και στάνταρ και τρίτον να βελτιώσουμε τη συμμόρφωση με τα εργασιακά πρότυπα και να επιβάλλουμε τη συμμόρφωση και τη θέση σε ισχύ των ε, νομικών διατάξεων και προβλέψεων. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα συνεργαστώ μαζί σας για να βρούμε συμβαστικές λύσεις, τροπολογίες, τις κανονιστικές διατάξεις, την νομική διατύπωση του κειμένου, για να πετύχουμε να σημειώσουμε πρόοδο σε αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Σάμιχ, παρακαλώ. Νομίζω ότι αναφερόμαστε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και χαίρομαι. Είναι μια οδηγία που θα πρέπει να την εξετάσουμε και το λέω διότι Πολλές φορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στα κράτη-μέλη δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση στην περιβόητη οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όλα αυτά είναι πολύ θετικά. Όμως δεν δίνεται αρκετή έμφαση στον αντίκτυπο που έχουν όλα αυτά στους εργαζομένους και στα δικαιώματά τους. Σε ορισμένες χώρες γίνεται αναφορά στην οικονομική ε, κατάσταση. Πώς αυτό όμως επηρεάζει τον εργαζόμενο και την ποιότητα ζωής του. Δίνεται, χρειάζεται να υπάρχει σαφήνεια στις συνθήκες εργασίας, στο πλαίσιο, στο περιεχόμενο αυτών. Καλό είναι ότι ε, έχουμε ψηφιακό φορμά. Όμως, ε, το καταλαβαίνει αυτό ο εργαζόμενος ή απλά κάποιος τσεκάρει ένα κουτάκι γιατί δεν υπάρχει καμία άλλη επιλογή να τσεκάρει. και η παράλληλη απασχόληση να την περιορίσουμε αυτή μόνο σε μια κατάσταση όπου υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και να σταματήσουμε εκεί. Αυτό είναι το λογικό για μένα. Απ' την άλλη όμως, να μην αναγκαστούμε να είμαστε σε μια κατάσταση που κάποιος κάνει ε, δύο, τρεις, τέσσερις δουλειές για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Και ποιο είναι ο αντίκτυπο στην εργασιακή ζωή και στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Ε, είναι θέμα ισορροπίας. Δηλαδή να είναι ενεργή αγορά ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Είναι πολύ λεπτό το σημείο ισορροπίας. Και τέλος, να γίνει αναφορά στην ανάγκη να μετρήσουμε όχι μόνο την οικονομική ανάπτυξη με τον αριθμό των νέων δουλειών που δημιουργούνται, αλλά να λάβουμε υπόψη μας π.χ. και τα ναι. νέα ημερομίσθια, τα νέα επίπεδα των μισθών. Και αυτά είναι σημαντικά. Όμως να έχουμε και ένα δείκτη για την ποιότητα της ζωής, γιατί τελικά πρέπει τις συνθήκες εργασίας να τις συνδέσουμε με τη διαφάνεια, με τη δυνατότητα να μπορούμε να μετρήσουμε την ποιότητα ζωής γενικότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω κάποιες αμφιβολίες για τον τρόπο με τον οποίο η συζήτηση αυτή ταιριάζει με το πεδίο αρμοδιότητας της Επιτροπής. Δεν είμαστε Επιτροπή για την απασχόληση και για τα εργασιακά. Εν πάση περιπτώσει θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Εάν όχι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδεχομένως να ε, θέλει να σχολιάσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ο εισηγητής μας έδωσε πάρα πολύ καλές εξηγήσεις για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να σας επιθυμίσω ότι η πρόταση αυτή έρχεται για να ανταποκριθεί στο πρόσφατο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στα ψηφίσματα του 2017 για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα ε, Κοινωνικών Δικαιωμάτων για τις συνθήκες εργασίας και την επισφαλή απασχόληση Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις συνθήκες εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τέλος, Υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια στις συνθήκες εργασίας, αλλά τίθεται και το θέμα της ποιότητας των συνθήκων εργασίας. Και γι' αυτό στην πρόταση έχουμε τα ελάχιστα δικαιώματα, μια σειρά ελάχιστων δικαιωμάτων που ε, ισχύουν για όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως του είδους της απασχόλησης. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η μήπως θέλει κάτι να προσθέσει. Από ό,τι βλέπω όχι. Επομένως προχωρούμε. Άρα ε, ε, ολοκληρώνουμε την εξέταση αυτού του ζητήματος στην ημερήσια διάταξη. Επομένω, σημείο 7 τη ημερησία διάταξη εξετάζεται και κλεισμένων των θυρών. Παρακαλώ, όσοι δεν δικαιούστε να παρίσταστε, ε, να αποχωρήσετε από την αίθουσα, γιατί τα επόμενα σημεία θα τα εξετάσουμε και κλεισμένων των θυρών.